πολιτικές ευαισθησίες συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην έκθεση. Με απόλυτη διαφάνεια και με το πνεύμα το οποίο ήταν ολονών μας όταν ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ την Επίτροπο Μάλστρομ για τον ενθουσιασμό της, για το, το birding sharing που θα ε, προσπαθήσει να παλέψει στο Συμβούλιο. Αν το παλέψει με τον ίδιο ενθουσιασμό πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Αν έπρεπε να σας δώσω μία περίληψη, μία σύνθεση των όσων υπόθηκαν, θα έλεγα όσο θα έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ του βορρά και του νότου αυτού του κόσμου, όσο θα υπάρχουν τέτοιες πολιτιακές διαφορές, όσο θα έχουμε τέτοιες τεράστιες διαφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, οποιαδήποτε πολιτική υποδοχή θα είναι αποτελεσματική και τμηματική. Εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε μια μεγάλη στρατηγική, μια πολιτική για την ανάπτυξη που θα βοηθήσει διαρθρωτικά στην κάλυψη των διαφορών μεταξύ Βορρά και Νότου. Όταν θα λύσουμε αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα θα λυθούν πιστεύω όλα αυτά και θα ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Όλοι κλωρώνεται η κοινή συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12. Τώρα, οι παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού ο κύριος Higgins. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύσει στην ε, μείωση, την ουσιαστική μείωση των ε, σοβαρών θανατηφόρων ε, τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε το 2033 ώστε να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Άδεια Οδήγησης. Τώρα έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Όμως, ε, ρεαλιστικά, τι αξίζει αυτό, τι αξία έχει. Ζητάμε από τους ε, χρήστες των δρόμων να ε, είναι αυτοί που θα προστατεύουν. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρώ ότι έχουμε την σύγχρονη τεχνολογία στη διάθεσή μας για να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, να επιταχύνουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν πρέπει να περιμένουμε παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μετζάρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η... Η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η χριστιανική πίστη είναι κοινέ ευρωπαϊκές αξίες που όλοι αναγνωρίζουμε. Ο, ο Γιώχαν Φανέστερχας έχει αναφέρει αυτές τις, ε, ε τις αξίες. Το, έχουν μαρτυρήσει το, το, το 42 ήταν ο μόνος ε, που καταδίκασε ε, τον, ε, την εκδίωξη των Εβραίων και αυτό είχε επιπτώσεις για τη Σλοβακία και την Ουγγαρία όπου η Γερμανή, ε, γερμανική μειονότητα εκδιώχθηκε. Είναι ε, ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα ακόμα υπάρχουν ενισχύ τέτοια πράγματα και σήμερα πρέπει ε, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να μαρτυρούν έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να

παστικοποιήθηκαν. Μιλάμε για τους ριζοσπάστες της Ουγγρικής μειονότητας. Και αυτό βέβαια και λόγω της αδιαλαξίας των Ουγγρικών αρχών. Κάθε φορά στις 15 Μαρτίου γίνεται, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται προκλήσεις, προβοκάτσιες εξ, Ούγγρων εξτρεμιστών που δεν δήλωσαν το άγαλμα ενός ήρωα της Επανάστασης του 1848. Παρακαλώ να μην γινόμαστε συνένοχοι. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκριζώσει το εθνικό μίσο σε μια περιοχή όπου τα προβλήματα του παρελθόντος πρέπει να επιληθούν από το ευρωπαϊκό πνεύμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μύρσκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Τι πιστεύετε είναι δυνατόν στο Βέλγιο, χάρη υπάρχει το ε, γαλλικό σχολείο, θα ήταν δυνατόν ε, στην ε, Γαλλία να κλείσει ένα γερμανικό σχολείο, αλλά στην Λετωνία όπου 40% είναι πληθυσμός ρωσόφωνος, αυτό είναι δυνατόν να κλείνουν τα σχολεία. Σήμερα στο Κοινοβούλιο της Λετωνίας ε, διάφοροι Ναζί θέλουν να οργανώσουν ένα δημοψήφισμα για το κλείσιμο των ρωσόφωνων σχολείων στην ε, Λετωνία και ταυτόχρονα έρχεται εδώ πολιτικός και λέει ότι είναι υπερήφανος ε, για την ενσωμάτωση στην Λετωνία τι θα γινόταν αν κλείσουν όλα τα ρωσικά σχολεία στην Λετωνία. Εγώ μπορώ να σας δώσω την απάντηση. Θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος στην ε, Λετωνία. Αν το Κοινοβούλιο δεν αντιδράσει σε αυτόν τον ρίζοσπαστισμό που εκφράζεται σήμερα στην Λετωνία, αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία δεν θα πρέπει να χειραγωγηθεί. Οι πολίτες θέλουν απαντήσεις και δράσεις. Θέλουν γρήγορα μέτρα, διαφανή μέτρα και να υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να κλείσουν τα πεπαλαιωμένα και προβληματικά εργοστάσια. Αντίστοιχα με αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογία της Φουκουσίμα. Παρακαλώ να κλείσουν στη χώρα των Βάσκων το πυρηνικό εργοστάσιο της Λαγκαρούνια γύρω από το οποίο κατοικούν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να υπάρξει πολεοδομική προστασία και πολιτική προστασία για να δούμε πού μπορούμε εμείς να, προστατεύσουμε αυτόν τον πληθυσμό σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής ούτως ώστε η εκένωση να γίνει τακτοποιημένα και γρήγορα. Η κυρία Άρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο... Ε, Ευρωπαίος Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι η ε, διάσωση των Ιρλανδικών τραπεζών δεν είναι βιώσιμη. Μιλάμε για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων ε, που ε, έχουν πληρώσει φόρους στην Ιρλανδία. 17 ε, δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος, για να μην αναφέρουμε και τα 200 εκατομμύρια ευρώ σε εκτακτή ανάγκη. Ένα μικρό νησί 4,4 εκατομμυρίων πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την τρέλα. Κάθε γυναίκα, άντρας και παιδί ε, έδωσε 160.000 ευρώ μόνο και μόνο για να διασώσει τις τράπεζες και χωρίς τους τόκους. Στην ε, Γαλλία 62 εκατομμύρια άνθρωποι ε, αν είχαν ταυτόσημη κρίση θα έπρεπε να δώσουν ένα 3 ευρώ. Αυτό θα ήταν δύσκολο αλλά βιώσιμο για την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κρίση του ευρώ, έχετε πει. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναγνωρίσει τι συμβαίνει και δεν αναγνωρίσει ότι ε, τα πράγματα είναι δύσκολα, τότε όχι μόνο το μέλλον της Ισλανδίας αλλά και της Ευρωζώνης θα είναι δύσκολο. Ο κύριος Τζουνκέρας. Καληνύχτα σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Καταλωνία στην τωρινή κρίση αντιμετωπίζει καλά, ε, θετικά μηνύματα. Έχει αυξήσει κατά 14% τις ε, εξαγωγές της, αλλά από την άλλη μεριά έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Το 40% ανεργίας των νέων. Η οικονομία της Καταλωνίας αποτελεί μοχλό για την Νότια Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να κάνει κάτι η Ευρώπη για αυτήν. Ο κύριος Βοτσακόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα στη Λιθουανία ένας νόμος για την παιδεία υιοθετήθηκε που αλλάζει το σύστημα το εκπαιδευτικό με τέτοιο τρόπο ώστε ε, πολλά σχολεία θα κλείσουν στην ε, Λιθουανία. Πρόκειται για διακρίσεις απέναντι στις ε, πολωνικές μειονότητες που ζουν στη Λιθουανία εδώ και πάρα πολλές γενές. Μετά τις οδηγίες να μην γράφονται πολωνικά ονόματα με τον πολωνικό τρόπο τιμωρήθηκαν ε, πολλοί διότι χρησιμοποιήσανε πολωνικά τοπονύμια. Έχουμε ένα άλλο, μια, έναν άλλο νόμο ε, που επιφέρει διακρίσεις στο σύστημα της παιδείας. Οι αρχές της Λιθουανίας δεν προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Έχουμε προβληματική κατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά όχι μόνο τη Λιθουανία, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τρενταφυλλίδη. Κυρία Πρόεδρε, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την έκθεση Όμεν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε πως στην έκθεση δεν υπάρχει ισορροπία και ότι ο ίδιος δεν θεωρεί ισορροπημένους αυτούς που την συνέταξαν. λίγες μέρες αργότερα τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές βροντοφώναζαν έξω από το ευρωκοινοβούλιο στις βρυξέλλες ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία δεν βρίζει μόνο τους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν την έκθεση της κυρίας Όμεν, αλλά και τους τουρκοκύπριους που σε ογκώδη συλλαλητήρια στην κατεχόμενη κύπρο διαμαρτύρονταν εναντίον της καταπίεσης που ασκεί πάνω τους η παρουσία 40.000 τουρκικού στρατού καθώς και ανυπολόγιστου αριθμού τούρκων επίκων. ο τουρκοκύπριος πολιτικός ιτζιάν μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε ότι η άγκυρα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο αλλάζει τη δημογραφική δομή ολοκληρωτικά με τη μεταφορά πληθυσμού από την τουρκία απειλώντα την ίδια την ύπαρξη τη τουρκοκυπριακή κοινότητα τονίζοντα ότι όποιο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω η ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί να αποδέχεται αυτή την παραβίαση. εμεί κυρία πρόεδρε ω κοινοβούλιο θα αποδεχθούμε αυτή την παραβίαση. σα καλώ όπω μεταφέρετε την πιο πάνω φωνή διαμαρτυρία των τουρκοκυπρίων τόσο στο συμβούλιο όσο και στην κομισιόν για να ενεργήσουν ανάλογα πριν είναι αργά. η Βόρεια Αφρική φλέγεται εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων σε Αίγυπτο, την Ισία, Λιβύη. Η κρίση αυτή συμπαρασύρει και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής με δυσμενή αποτελέσματα πολιτικά αμφίβολα και αόριστα. Δεύτερον, παράλληλα υπάρχει σημαντική αυτονόμηση της τουρκίας από τα κέντρα αποφάσεων της δύσης με τη σύγκρουση της άγκυρας με το ισραήλ τη σύσφιξη σχέσεων τουρκίας ιράν βραζιλίας. η τουρκία αυτονομείται τόσο από τις αμερικανικές πολιτικές για τη μέση ανατολή αλλά και από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για μελλοντική ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση. η αστάθεια εξακολουθεί να υπάρχει στις χώρες της πρώην ιουγκοσλαβίας και τροφοδοτεί εθνικιστικούς κύκλους τέλος ασφαλείς διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι το 2030 τριάντα οι μοαμεθενικοί πληθυσμοί που σήμερα ανέρχονται σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια δισεκατομμύρια θα είναι 2,2 δισεκατομμύρια ενώ οι ευρωπαίοι θα απομειωθούν τουλάχιστον κατά 50 εκατομμύρια κατοίκους. ερωτάτε καταλαβαίνουν οι ηγέτες της ευρώπης ότι η αποσταθεροποίηση του νότου θα έχει επιπτώσεις δυσμενείς όχι μόνο στο ευρώ αλλά και στη γεωπολιτική σταθερότητα του δυτικού συστήματος ασφαλείας. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. κύριος Η κυρία Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις της οικονομικής ε, κρίσης στην Ιρλανδία, στην οικονομία στην Ιρλανδία, όμως ε, με μεγάλη μου θλίψη ενημερώθηκα για το φόνο ενός ε, μέλους της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Ρόμαν Κέρ, 25 ετών, πέθανε στα χέρια τρομοκρατών ε, το Σάββατο το απόγευμα. Ήταν ένας καθολικός αστυνομικός ε, και φωνεύτηκε όταν ξεράγει βόμβα κάτω από το αυτοκίνητό του καθώς έφευγε από τη δουλειά του το Σάββατο. Πέθανε επί τόπου. Θα ήθελα να καταδικάσω αυτή τη φρικαλαιότητα και να ζητήσω στο μέλλον αυτές ε, οι βίες πράξεις τρομοκρατών αντί να φέρουν την Ιρλανδία πίσω στο σκοτεινό της παρελθόν ε, να ε, δυναμώσουν την πολιτική διαδικασία. Έχουν ως τώρα το τελευταίο διάστημα εφητευτεί χιλιάδες τέτοιες βόμβες κάτω από τα αυτοκίνητα των αστυνομικών και πολλές από αυτές δεν εξεράγησαν ευτυχώς. Ελπίζω ε, όλες οι πληροφορίες ε, αυτές που αφορούν στο φόνο να δοθούν στην ε, αστυνομία και να κάνουμε όλοι μαζί έκκληση γι' αυτό. Πρέπει να μάθουμε τα πάντα γι' αυτόν τον φρικτό φόνο έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι δράσεις και να μην προστατευτούν. Πρέπει αυτό να γίνει για το μέλλον της χώρας μας και για το σεβασμό ενός γενναίου αστυνομικού και της πενθούσας μητέρας του και οικογένειάς του με λυπεί το ότι δεν σεβάστηκαν την ομιλία αυτή πολλά μέλη αυτού του κοινοβουλίου. Ο κύριος Πουπάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την επικύρωση της σύμβαση στο ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα 27 κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση και ίσες δυνατότητες επιλογών, διασφαλίζοντα σε αυτούς τους συμπολίτες μας πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Όμως, όπως διαπιστώνετε αυτό δεν ισχύει για όλους. γύρω στα 30 εκατομμύρια τυφλοί που ζουν στην ευρώπη ακόμα και για τις καθημερινές τους δραστηριότητες όπως η αγορά προϊόντων αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες αφού για να μάθουν τι περιέχει μια συσκευασία πρέπει πρώτα πάντα να στηρίζονται στους άλλους. θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την επιτροπή να προβεί σε ευρία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας συσκευασίε των προϊόντων σε γραφή braille και συγχρόνω να καλέσω του συναδέλφους μου εδώ μέσα να στηρίξουν με την υπογραφή τους τη γραπτή δήλωση 14. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής προκάλεσαν κάθε άλλο καθησυχασμό η σαφής πρόβλεψη δυνατότητας κράτους μέλους να προβεί σε αναδιάρθρωση χρέους μετά το 2013 αποτελεί ξεκάθαρη υπαναχώρηση από την αρχική θέση της ευρωπαϊκής ένωσης όταν ξέσπασε η κρίση ότι δηλαδή η αναδιάρθρωση χρέους θα αποκλειστεί με κάθε κόστος. και ήδη στην ελλάδα και πάλι ανακοινείται η σχετική συζήτηση από διακεκριμένους οικονομολόγους σε διεθνές επίπεδο και από τις αγορές. τι συνέβη λοιπόν και άλλαξε αυτή η στάση; καταβλήθηκε κάθε κόστος κάθε προσπάθεια; μήπως τελικά εξαντληθήκαμε; η αλήθεια είναι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει. η ύφεση βαθαίνει στην ελλάδα αντί να ανακόπτεται και το θλιβερότερο η ε, τα κρατικά έσοδα είναι στο μείον 9% το πρώτο δίμηνο όταν έπρεπε να είναι στο συν οκτώ με βάση το μνημόνιο για το 2011 και το θλιβερότερο η ανεργία ήδη ξεπερνάει το 15%. Σε αυτά η απάντηση είναι μία. Ανάπτυξη. Τη βλέπουμε όμως αυτήν την ανάπτυξη. Όχι. Αναπτυξιακές πολιτικές χρειαζόμαστε, όχι αναδιπλώσεις και συζητήσεις για αναδιαρθρώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Προεδρία του Ουγγρικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή ε, κάνει μια ενδιάμεση ε, αξιολόγηση. Ε, έχει ψηφιστεί το έκτο πακέτο στο Συμβούλιο. Μιλάει για την ανταγωνιστικότητα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Φεβρουάριο στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε μια μεγάλη τομή για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Στην Επιτροπή Συνοχή στην γεωργική πολιτική ε, έγιναν ε, βήματα, όμως υπάρχουν και ανοιχτά ε, θέματα όπως η στρατηγική για τους Ρωμά. Με την ψήφιση αυτής της στρατηγικής η Ευρώπη ανέφερε την υποχρέωσή της για υποστήριξη των Ρωμά. Ε, ελπίζω και εσείς να ε, υποστηρίζετε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κύριε Άντρα. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, κυρία Ντότς ήθελα να μιλήσω για την οικονομία. Αλλά νομίζω ότι στην Βόρειο Ιρλανδία η δολοφονία ενός καθολικού ιερέα άλλαξε την κατάσταση. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η τραγωδία για την Ιρλανδία και για την οικογένεια που επλήγει. Είχε τελειώσει την αρχική εκπαίδευση το Δεκέμβριο, ήταν 25 ετών και μια βόμβα εξεράγει μπροστά στο αυτοκίνητό του. Χτες ήταν η ημέρα ε, των μητέρων ε, και είπε ότι δεν θα έπρεπε ε, να αποθαρρυνθούν οι καθολικοί να διαδηλώσουν έκανε έκκληση σε όλους τους καθολικούς να μην αποθαρρύνονται από αυτήν την δολοφονία θα έπρεπε να προσπαθούν να επιτύχουν την ισότητα. Είπε μέσα στη λύπη της δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στις ζωφερές ημέρες του τρόμου. Ήμασταν τόσο υπερήφανοι για τον γιο μας. Δεν θέλουμε ο θάνατός του να είναι μάταιος, να είναι επιματέο. Θα πρέπει όσοι διέπραξαν αυτήν την δολοφονία ε, να έρθουν ε, να ομολογήσουν ε, και είναι καθήκον μας να εξακολουθήσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας. Ο αξιότιμος Ήβαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, στη Ρουμανία έχουμε ένα νόμο που λέει ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει να έχουν μεγαλύτερους μισθούς γιατί σήμερα οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί. Δηλαδή το δικαστήριο δικαίωσε τους ε, καθηγητές και τους δασκάλους για την αύξηση του μισθού τους <laughs> αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να εφαρμόσει τον νόμο. Και προτείνει ένα νέο νόμο που περιορίζει τους μισθούς των δάσκαλων και καθηγητών. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Και επίσης πλήττονται βασικοί στόχοι της, ε, της Ευρώπης 2020 η οποία στοιχηματίζει ιδιαίτερα στην παιδεία. Χρειαζόμαστε καλοπληρωμένους δασκάλους για να έχουμε αποτελεσματική παιδεία. Ο κύριος Θανασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από την καταστρεπτική πολιτική του καθεστώτος Μπασέσκου Μποκ, Το σύστημα υγείας της Ρουμανίας έχει φτάσει σε πτώχευση. Τα νοσοκομεία έχουν τα χάλια τους και το υγειονομικό προσωπικό βρίσκεται σε κατάσταση ανέχειας. Τα προβλήματα δεν λαμβάνονται υπόψη από την τωρινή κυβέρνηση. Οι παθολόγοι έχουν ε, φτιάξει έναν σύλλογο και για να μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα με την κυβέρνηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας τα λέω όλα αυτά διότι άμα αποτύχουν τότε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι το κράτος πλέον δεν υπάρχει. Ο κύριος Μασίπ. Ο Φίλιππος ο των Βουρβώνων, ο οποίος είναι πρίγκιπας της Αστούριας, που είναι η εκλογική μου περιφέρεια, υποδέχτηκε τον πρίγκιπα ε, Κάρολο της προάλλες. Και όλα αυτά βαίνουν σε καλές και με καλές σχέσεις, αλλά σήμερα που έχουμε δημοκρατία δεν μπορούμε εμείς να δεχόμαστε την κατοχή του Γιβλαρτάρ από τους Άγγλους. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με την Βόρεια Κύπρο. Εγώ μιλάω τώρα για το Γιβλαρτάρ που το επισκέφτηκα πρόσφατα. Ο κύριος Φαγιόν δεν είναι εδώ. Η κυρία Φαγιόν. Η κυρία Νευρεδάλοβα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βελτιώσει την αγωνιστικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Το μέλλον είναι η νεολαία μας και η εκπαίδευσή της. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκεται σε μια θέση που η παιδεία δεν έχει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Υπάρχει κρίση και οι επιπτώσεις της σήμερα έχουν να κάνουν και με αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε το οικονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο θα θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη δεν ε, δίνουν ε, κονδύλια για αυτό το θέμα ε, γιατί ε, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αν θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Ο κύριος Τρεμόσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να καταδικάσω ε, την επίθεση στην εσωτερική αγορά και την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των ανθρώπων και των αγαθών έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες καταλωνικές ε, ε, εφημερίδες ενημέρωσαν ότι Γάλλοι αγρότες κατέστρεψαν προϊόντα Αυτές οι επιθέσεις ως τώρα έχουν επαναληφθεί άλλες δύο φορές από την αρχή του έτους, το 2011. Η τελευταία συνέβη πριν από μερικές εβδομάδες όταν κάποιοι επικετοφόροι σταμάτησαν άλλο ένα ε, φορτηγό από την Καταλωνία, επιτέθηκαν στον ε, οδηγό και έριξαν δίζελ πάνω σε 20.000 κιλά ε, κρέατος. Αυτή λοιπόν η καταστροφή των προϊόντων που έρχονται εκτός της Γαλλίας έχει επίπτωση στην ε, ε κρέατοβιομηχανία των ε, Καταλωνίας. Έχουν πέσει κατά 50% οι πωλήσει. Έχω καταθέσει ένα γραπτό, ένα γραπτό ερώτημα ε, στην Κομισιόν, ε, ελπίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει αυτή την απαράδεκτη επίθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βαντίμ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σόγκορ. η πολιτισμική ε, οι πολιτισμικές διαφορές είναι μία από τις αξίες της Ευρώπης και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τη διατηρήσουμε. Στην Ήπειρό μας υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι ε, και πολιτιστικές αξίες που ε, βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Οι τσάνγκος που ζουν στην Ρουμανία είναι μία τέτοια μειονότητα. Η σύσταση 1521 ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μειονότητα των Τσάγκο. Ε, κάποια πράγματα τα έχει ήδη υιοθετήσει η ρουμανική κυβέρνηση όμως ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει από τα κόμματα να δώσουν λογαριασμό έτσι ώστε ε, να δούμε γιατί λειτουργεί έτσι αυτή η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως τώρα δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Λοιπόν, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τιμηθεί η αρχή ε, της των πολιτισμικών διαφορών που βρίσκεται στην παραγραφό 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης θα πρέπει να κάνει τα πάντα των ε, Μολδαβών Ούγκρων Τσάγκος. Ε, Τελευταία τοποθέτηση η κυρία Εστάρας. Τον προηγούμενο Ιανουάριο η Κομισιόν ενέκρινε τη στρατηγική για, την, ε, για να καταπολεμήσει την πρόορη εγκατάλειψη του, του σχολείου. Και αυτό εν ώψη της στρατηγικής 2020 θέλει να μειώσει κατά 10%, κάτω από το 10% αυτό το ποσοστό. Δεν γίνεται όμως αναφορά στην ανικανότητα και σε αυτό το λεπτό θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το θέμα γιατί στις 4 Μαΐου στις Βρυξέλλες θα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Παιδείας για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της ανικανότητας της αναπηρίας ε, πνευματικής αναπηρίας σε αυτόν τον τομέα που χρειάζεται ειδική παρακολούθηση και συνεχή ε, κατάρτιση για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην αγορή εργασίας. Το άρθρο 24 της χάρτας του ΟΙΕ το προβλέπει ούτως ώστε να μην αποκλείονται αυτά τα άτομα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα, έκθεση της κυρίας Γέγλε ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές. Για τέσσερα λεπτά η κυρία Γέγελ.